Ε, πρώτο μέρος των ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Ε, η πρώτη ερώτηση έχει υποβληθεί από τον κύριο Παπαστάμκο. Ε, κύριε Μπαρνιέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαστάμκο για αυτή την ερώτηση που αφορά ένα θέμα το οποίο επειδή είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου θεωρείται πρωταρχικής σημασίας. Η... Τα Ιδρύματα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ε, παίζουν σημαντικό ρόλο και σε περίοδο κρίσης όπως τώρα δείχνει ότι η λειτουργία τους έθεσε και θέτει κάποια προβλήματα με επιπτώσεις πολλές φορές οι οποίες είναι πολλές φορές επαχθείς. Γι' αυτό το λόγο το G20 έλαβε σωστά την απόφαση να δημιουργήσει ένα όργανο εποπτείας και να θεσπίσει κανόνες κυβέρνηση. Θα ήθελα να σας ότι στη στιγμή της κρίσης η Κομισιό πάρα πολύ γρήγορα επί αυτού του θέματος επομίστηκε τις ευθύνες της και έκανε θέμα προτεραιότητα το θέμα λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων. Από τον Σεπτέμβριο του 2009, ένα χρόνο μετά την ε, χρεοκοπία τη Λέμμαν, εγκρίθηκαν κάποιοι κανόνες την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να ποτίσω φόρο φινή στην εργασία την οποία έκανε ο κ. Κόζε, ιδιαίτερω ο εισηγητής, για να ανταποκριθεί στο πρόβλημα το οποίο ήταν ο τρόπο λειτουργία αυτών των ε, ιδρυμάτων και που συνεισέφεραν σοβαρά στην ε, ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση καταγραφής όλων των ε, ιδρυμάτων αυτών πιστοληπτική, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητες. Αυτό γίνεται πρώτα απ' όλα για να σταματήσουν ε, οι διαφορές προάσπισης συμφερόντων για να δούμε πώς γίνεται σωστά η αξιολόγηση και για να μπορούν αυτά τα ιδρύματα να ενεργούν με διαφάνεια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Έχω εμπιστοσύνη ότι αυτοί οι νέοι κανόνε των Ιδρυμάτων αυτών θα βελτιώσουν με αποφασιστικό τρόπο την ανεξαρτησία και την ακαιρεότητα τη όλη διαδικασία αξιολόγηση, θα βελτιώσουν τη διαφάνεια όλων αυτών των δραστηριοτήτων και την ποιότητά του, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν ε, τα χρέη ε, των επισήμων κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα, κύριε Παπαστάμκο, όσον αφορά την δημιουργία μιας ε, δημόσιας Ευρωπαϊκής Αρχής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στα πλαίσια των ελεκτικών λύσεων που έχουμε για το παρόν σύστημα. Μια τέτοια ιδέα, μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να αξιολογηθεί με σοβαρότητα, κυρίως όσον αφορά το θέμα της ευθύνης θα πρέπει λοιπόν να σας πω με σαφήνεια κύριε Παπαστάμπτο ότι αυτό το οποίο θέλουμε κυρίω είναι να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κανονισμό του 2001 και να μπορεί το ανανεωμένο παρόν σύστημα να λειτουργεί σωστά. Δεν κλείνω όμω την πόρτα στην ιδέα αυτή την οποία παρουσιάζεται για τη δημιουργία και την σύσταση μια Ευρωπαϊκή Αρχή, θα πρέπει να δούμε το όλο θέμα κάνοντα την αξιολόγηση του κανονισμού του 2009 προβλέπεται η αξιολόγηση στον ίδιο τον κανονισμό εξάλλου και η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την αξιολόγηση που θα κάνει ως τον Δεκέμβριο του 2012. Αυτό το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα προτείνει η Επιτροπή μελλοντικά να γίνει και αλλαγή του κανονισμού αυτών των Ιδρυμάτων ώστε να έχει η Ευρωπαϊκή Αρχή την πλήρη εποπτεία της αξιολόγησης τους. Το ζητήσατε εσείς και το ζήτησαν και οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων που συμφώνησαν με αυτή την αρχή. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το οποίο λέγεται η μεταφορά σε αυτή την νέα η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή ε, ελέγχου αυτών των Ιδρυμάτων Αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο θα συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επίτροπο κύριο Μπαρνέ για την ε, απάντησή του και θέλω να σας πω κύριε επίτροπε ότι είναι ένα θέμα για το οποίο άσκησα κατ' επανάληψη κοινοβουλευτικό έλεγχο ήδη από το 2006 πολύ πριν εμφανιστεί η διεθνής οικονομική κρίση. Υπάρχουν δύο παράδοξα κατά τη γνώμη μου. Υφίστανται διεθνοποιημένοι οίκοι αξιολόγησης χωρίς διεθνοποιημένη εποπτεία. Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι ιδιωτικά σχήματα και συμφέροντα εκτός Ευρώπης εμφανίζονται επικυρίαρχα έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών. θα ήθελα κύριε επίτροπε και απευθύνω ε, ε, έκκληση να κινηθεί η επιτροπή με πιο γρήγορο ρυθμιστικό χρόνο με πιο γρήγορο ρυθμιστικό βήμα. και τέλος ποια είναι η γεωγραφική έδρα και πώς κατανέμεται ο κύκλος εργασιών αυτών των οίκων αξιολόγησης. σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κύριε Παπαστανκό, ξέρω. Εδώ και πόσο καιρό ασχολείστε τόσο σοβαρά με το θέμα. Το ξέρω και σήμερα. Γίνεται αυτή η συζήτηση πρώτη φορά μεταξύ μας. Λαμβάνω υπόψη το νέο κανονισμό που πρότεινε και η προηγούμενη επιτροπή από τον κύριο Μπαρόζο που βελτιώνει τα πράγματα και θέτει νέες απαιτήσει για αυτούς τους οίκους. Η τελευταία πρόοδος θα επιτευχθεί, στην πρόταση θα σας κάνω, σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες, είναι ότι θα υπάρχει από τη ΣΜΑ μία εποπτεία. Και σωστά λέτε ότι δεν είναι ο πρώτος, το μόνο θέμα όπου σε μία ενιαία αγορά και ολοκληρωμένη αγορά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, κάποια σχήματα όπως λέτε και εσείς που ενεργούν. Υπενθυμίζω κύριε Παπαστάμκο ότι στις μισές χώρες ο μικός, μισός τραπεζικός αν θέλετε τομέας ανήκει σε αλλοδαπές τράπεζες. Και το θέμα της εποπτείας παρόλα αυτά παραμένει εθνικό θέμα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλή δουλειά ολοκλήρωσης και ανισομάνωτη. Και στα πλαίσια των νέων καθηκόντων που θα δοθεί στην ΣΜΑ θα υπάρχει αυτή η εποπτεία ευρωπαϊκή όπως την επιθυμείτε εσείς. Τώρα, όσον αφορά τη χώρα σας, η οποία πραγματικά τραντάχθηκε από τα τελευταία γεγονότα, θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Δεν θα κάνω καμία παρατήρηση για το τι ακριβώς έγινε. Θα πρέπει ούτως ή άλλως όταν αυτή η οίκη αποφαίνονται για κάποιες χώρες να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κυρίαρχη χώρα και βεβαίως το θέμα του χρέους είναι κάτι που απασχολεί τους πάντες, όλους τους φορολογούμενους και όλο τον πληθυσμό. Το Σάββατο, Υπουργείο Οικονομικών και ε, στη Μαδρίτη είπαν οι Υπουργοί ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέρη ώστε να μην χρειάζεται οι φορολογούμενοι να βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Και βεβαίω ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν αυτοί οι οίκοι και μπορούν να επηρεάσουν τους επενδυτές είναι γνωστό σε όλου. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βάλουμε υψηλά τον πύχη πρώτα απ' όλα να επαγρυπνούμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και θα ε, κάνω προτάσεις ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εποπτεία όσον αφορά τη λειτουργία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την εξαιρετική ε, έκθεση ε, νομίζω μπορεί να μας κάνει αισιόδοξου όσον αφορά την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Αξιολόγησης Πιστοποιητικής Ικανότητας για να είμαστε ανεξάρτητοι από ε, ιδιωτικούς οίκους αξιολόγησης. Εμένα με ενδιαφέρει εδώ πέρα όχι η έδρα, ε, θα μας ενδιαφέρει βέβαια στη συνέχεια πώς η, αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή αντικειμενικά αλλά και ως προς τη δομή της θα λειτουργεί. Και θέλουμε να είναι ένα ισχυρό όργανο και θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες διαδικασίες προβλέπονται, τι συνέπειες ε, θα, έχει, ε, θα υπάρχουν σε περίπτωση που διαπιστωθεί αρνητική πιστοληπτική ικανότητα. Euh, Κύριε βουλευτά, ο κύριος Παπαστάμκον μου έκανε το ρίο του κατά πόσον θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή ως δημόσια αρχή από ό,τι κατάλαβα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητα. Εγώ δεν μπορώ να πάρω δεν ξέρω που θα κατευθυνθεί η Κομισιό, διότι η πρόταση Κομισιό αφορούσε την ανανέωση του παρόντος συστήματος που διέπει τα ιδιωτικά αυτά σχήματα αξιολόγησης και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια ώστε να μην υπάρχουν επικαλυπτόμενα συμφέροντα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έχουμε αυτό τον κανονισμό ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και θα συμπληρώσουμε την όλη δράση μας με τον ρόλο εποπτείας που θα αναθέσουμε στη ΣΜΑ, σε αυτή την νέα Ευρωπαϊκή Αρχή, όπως το επιθυμεί και ο κύριος Παπαστάμκους. Είπα, δεν έκλεισα την πόρτα, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε αυτό το business model ε, ε, πώς θα λειτουργήσει. Πρόκειται για μια ιδέα ενδιαφέρουσα την οποία όμως θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, δεν το ξέρω ακόμη. Και βεβαίως εδώ πρέπει να τεθεί το θέμα της παρέμβασης των δημοσίων αρχών. Και εάν υπάρχει μια δημόσια τέτοια ευρωπαϊκή αρχή θα πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα αντικρωμένων συμφερόντων. Αλλά ειλικρινά πρέπει να πω ότι για να δουλέψουμε σοβαρά και για να μην αυτοσχεδιάζουμε θα πρέπει να έχουμε χρόνο για να μπορέσουμε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις που θα αφορούν τη θέσπιση αυτού του οργανισμού και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν αφού τα έχουμε μελετήσει προσεκτικά. Ευχαριστώ. Ε, ο κανόνας είναι ότι όταν κάποιος ε, συνάδελφος δεν είναι στην αίθουσα κατά τη συζήτηση ερώτησή του, η ερώτηση καταπίπτει. Αλλά εξαιτία των εξαιρετικών περιστάσεων αυτής της Ολομέλειας, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι, θα αναγνώσω τα ονόματα όσων δεν είναι παρόντες και θα λάβουν υπό αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις μια γραπτή απάντηση στο ερώτημά τους. Αλλά δεν θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια. Ε, αυτοί λοιπόν που θα πάρουν αυτή η απάντηση, αλλά δεν είναι εδώ στη σειρά που έχουν υποβληθεί ερωτήσει ε, Είναι ο κύριος ε, Μπαλτσίτης, ο κύριος ή η κυρία ε, Νάιτε, και η επόμενη ερώτηση προς τον κύριο Αλμούνια που αφορά ερωτήσεις προς επιτρόπους που έχουν οριστεί για αυτή τη σύνοδο είναι από τον κύριο Άλουαρντ. Ε, οπότε σε αυτήν την ερώτηση, την ερώτηση 28, παρακαλώ τον κύριο Επίτροπο για την απάντησή του. επομένως, μόλις έρθει ο κύριος Σαλμούνια, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την απάντηση. Συνεχίζω τώρα με τους ερωτώντες που δεν είναι παρόντες. Ο κύριος Στούσας θα λάβει και αυτός γραπτή απάντηση. Ο κύριος Κρόλη, ο κύριος Ζιόμπρο και η επόμενη ερώτηση Οκ. Αλλά μπορούμε, είναι ο Επίτροπος ο κύριος Ντεούτ είναι εδώ. Yes. Ωραία. Οπότε μπορούμε τώρα που Mr. welcome. Are you, are you, are you ready to... Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμος να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Έλουαρτ. Ωραία. Έχετε λοιπόν το λόγο για να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Έλουαρτ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, ήμουνα στην πόρτα της αιθούσης. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τι εξελίξει όσον αφορά τα έξυπνα τηλέφωνα και τι σχετικέ αγορέ, όπω αναγνωρίζει και ο κύριος Βουλευτή στην ερώτησή του, σε ορισμένε περιπτώσει έχουν δημιουργηθεί νέε αγορέ. Η Κομισιόν είναι απόλυτα δεσμευμένη στο να διασφαλίσει ότι οι αρχέ τη Ένωση ε, περί ανταγωνισμού θα γίνονται σεβαστές, λαμβάνοντα υπόψη βέβαια τη δυναμική τη αγορά αυτή. Σε πρόσφατε περιπτώσει όπω η Microsoft και η Intel έδειξαν, ε, η Κομισιόν λαμβάνει κάνει ενισχυμένη δράση ώστε να διασφαλίσει ε, ότι οι κανόνες ανταγωνισμού θα επιτρέψουν στους καταναλωτέ να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορε επιλογέ και τι τεχνικέ εξελίξει και την καινοτομία ε, αναγνωρίζουμε ότι η τεχνολογία είναι στην καρδιά της επιτυχίας της Ευρώπης στις ε, τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας δεύτερης και τρίτης γενιάς. ταυτόχρονα γνωρίζει τις εξαιρετικές τεχνικές εξελίξεις, εξελίξεις που οφείλονται σε ε, νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες ψηφιακές. Η αγορά είναι αυτή που θα επιλέξει βέβαια τον νικητή, αλλά η Κομισιόν ε, τονίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας και τις, ε, το ανταγωνισμό ανάμεσα στις τεχνολογίες διαφόρων ε, ε, εταιριών και βοηθά στην να αποφευχθεί το μονοπόλιο καθώς και οι κυρίαρχες θέσεις ανάμεσα σε γειτονικέ αγορές. Οι ανοιχτές πλατφόρμες εξυπηρετούν αυτό το στόχο και επιτρέπουν τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών επιπλέον των συστημάτων software. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλγουαρντ έχει το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την απάντησή τη να αλλάξω ελαφρώ, γιατί υπήρξαν διάφορε νέε υποθέσει που αφορούν την έννοια της ε, λογοκρισίας ε, επί του περιεχομένου, που είναι ε, επαναλαμβανόμενη σε αυτή την τεχνολογία. Ορισμένε εφαρμογέ έχουν αποκλειστεί από ορισμένου κατασκευαστέ λόγω του περιεχομένου τους. Η Κομισιόν μπορεί να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει αυξανόμενο ανταγωνισμός στην πρόσβαση της πληροφορίας, της πληροφορίας μέσω της νέας τεχνολογίας και ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα επιλογής. Yes, indeed, I, I, know that uh, The elements included in your second question. Γνωρίζω ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δεύτερη ερώτησή σας και το θέμα που μόλι δείξατε μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ανταγωνισμού στην αγορά. Παρακολουθούμε στενά διαρκώ το θέμα. Δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένε ε, έρευνες, αλλά έχουμε στοιχεία στα χέρια μας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα προβλήματα τα οποία εσείς παρουσιάζετε και ανησυχίε σας είναι υπαρκτά και είναι ρόλος μου και ρόλος μας ως αρχή επί του ανταγωνισμού να αποφύγουμε το είδος κυρίαρχης θέσης για κομμάτια της αγοράς, για τις νέες εισόδους και εν τέλει να προωθήσουμε την πρόοδο για τους καταναλωτές, για αυτές τις νέες τεχνολογίες, ώστε να ωφελούνται και όχι να υποφέρουν από τις εξελίξεις και τις βελτιώσεις των τεχνολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Η πρώτη από τον κύριο Ρούμπικ για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στον κανονισμό Ρώμη 1 ε, έχουμε ρύθμιση για την ανταλλαγή δεδομένων ε, και για τις ε, τηλεφωνικές συνομιλίες. Κάθε πάροχος υπηρεσιών στην Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε πελάτη. Ε, κάποιοι όμως ε, δεν είναι διατεθειμένοι να ε, παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη. Πιστεύετε εδώ ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι εθνικές αρχές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που η Κομισιόν αναφέρεται στην πτυχή της ανταγωνιστικότητας στο θέμα αυτό. Η ερώτησή μου είναι αν υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις, ανάλογες υποθέσεις ε, του ΔΕΚ και μπορούν αυτές ε, να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση όσον αφορά την ε, πρόσβαση και έχουμε περιπτώσεις καταναλωτών που έχουν προσφύγει κατά των παρόχων υπηρεσιών. Κύριε Αλμούνια, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τις ερωτήσεις σας πιστεύω πως θα πρέπει να συνδυάσουμε έναν κατάλληλο κανονισμό και τα μέσα ανταγωνισμού. Για ορισμένες από τις πτυχές που θίξατε στις ερωτήσεις και στην παρέμβασή σας, τα όργανα περί ανταγωνισμού, τα μέσα, τα εργαλεία μάλλον που αφορούν τον ανταγωνισμό έχουν, έχουν δουλέψει, έχουν λειτουργήσει, αλλά δεν αποκλείεται ότι όταν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουμε τις ρυθμιστικές μας ε, ε, αρμοδιότητες. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και θα το ξαναπράξουμε όταν και όπου αυτό χρειαστεί ε, νομίζω πως τα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, παραπληρωματικά. Όσον αφορά τη δική σας ερώτηση, με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαι δυναμικός, δεν γνωρίζω ε, ποια είναι, ποιες είναι οι καταγγελίες των μεμονωμένων πολιτών ενώπιον των δικαστηρίων. Έχουμε λάβει, λαμβάνουμε μάλλον κάποιες πληροφορίες, ορισμένες φορές και ε, καταγγελίες και κάθε φορά που χρειάζεται να αντιδράσουμε γιατί θεωρούμε πως οι πληροφορίες που λάβαμε ή οι καταγγελίες που στέλνονται στην Επιτροπή πρέπει να να λάβουν απάντηση από την πλευρά μας, ε, το κάνουμε, απαντούμε. όπως είπα και στην προηγούμενη μου απάντηση, σε αυτό το τομέα, σε αυτό το τομέα, με όλα αυτά τα προβλήματα, ασχολούμαστε με κάποιες έρευνε που δεν μπορώ δημόσια να σας αναφέρω γιατί λόγω της φύσης τους πρέπει να είμαι διακριτικός. Ευχαριστώ. Ο Ρωτών, κύριος Τούσας, ε, θα λάβει γραπτή απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο Αλμούνια. Οι επόμενες ερωτήσει είναι για την ε, Επίτροπο Νέλη Κρός, η οποία όμως δεν νομίζω ότι είναι εδώ ακόμα. She's not here yet, correct? Okay. Δεν είναι εδώ ακόμα, κύριε Κρούς, σωστά. Ε, από ε, τον, ε, τον κύριο Άιλαρντ, αλλά θα πρέπει να περιμένετε όμως αυτή η κυρία Κρούς. Γραπτές απαντήσεις θα λάβουν ο κύριος Γιόμπρο, η επόμενη ερώτηση προς τον Επίτροπο Τεγκούτ είναι από τον κύριο Χουντή. είναι η ερώτηση 32. Ε, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για την απάντηση. Thank you, uh, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε από τον τραπεζικό τομέα, αλλά από τον δημόσιο τομέα. Ο τραπεζικός η έλλειψη σταθερότητας ε, ε, του τραπεζικού συστήματος ε, όμως έχει αυξηθεί λόγω της έκθεσης των τραπεζών στα δημόσια ομόλογα. Η Κομισιόν αναλύει μόνη της την ελληνική οικονομία και την οικονομική κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλές πηγές ε, πληροφόρησης, μεταξύ άλλων ε, τους οίκους αξιολόγησης. Και η Κομισιόν εξετάζει την εφαρμογή των ε, πρόσθετων μέτρων που ανακοινώθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στις 31 Μαρτίου του 2010 με στόχο την επίτευξη των στόχων της Κομισιόν του 2010 το 8% ε, του ενεργητικού των τραπεζών ε, έχουν τη μορφή ομολόγων ε, κρατικών και αναμένεται να φτάσουν στο 8% το 2010 λόγω της ασθενούς οικονομίας τράπεζες ε, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, εφόσον έχουν αποκλειστεί από τις ε, διεθνεί χρηματαγορές. Η Κομισιόν αναλαμβάνει την ευθύνη τη για να διασφαλίσει την μακροοικονομική σταθερότητα στην, στη ζώνη του ευρώ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η Γαλλία και η Γερμανία είναι οι χώρε που ανησυχούν περισσότερο όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα. Η έκθεσή του δεν είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά το ΑΕΠ. Ε, είναι αρκετά σημαντικέ όσον αφορά του ισολογισμού ε, των μεμονωμένων τραπεζών. Ε, το 10% των ελληνικών τραπεζών επενδύουν στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την απάντηση ε, προφανώς υπάρχουν προβλήματα στις τράπεζες στην ελλάδα υπάρχει αυτή η ρευστότητα που έχει παρέξει και το ελληνικό δημόσιο η οποία δυστυχώς δεν πάει προς την πραγματική οικονομία αλλά η επισήμανση που θα ήθελα να σας κάνω είναι κάθε φορά που βγαίνει ε, η ελλάδα ανακοινώνει κάποια μέτρα ανακοινώνονται κάποιες ε, μορφές δανεισμού βγαίνουν αυτοί οι περίφημοι οίκοι αξιολόγησης χαμηλώνουν την πιστοληπτική ικανότητα της ελλάδας και των ελληνικών τραπεζών είναι θλιβερός αυτός ο ρόλος. έγινε και λίγο κουβέντα και δεν θέλω να την ανακυκλώσω. είναι πράγματι αναξιόπιστη αυτή η οίκη αξιολόγηση. είναι αμερικάνικες ιδιωτικές εταιρείες. είναι απαράδεκτο να τους αποδέχεται η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ακόμα και σήμερα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ως αξιολογητές. το ερώτημα που τίθεται και ακούστηκαν πριν οι απαντήσει. εντάξει το 2013 πιθανόν να ρυθμιστεί. Τώρα άμεσα είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί να μην λαμβάνουν υπόψη τι αξιολογήσει αυτών των οίκων. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όπως μόλις είπα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις, στις αναλύσεις της τα στοιχεία που έχει από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητα, αλλά και τις δικές της αναλύσεις. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά το τι γίνεται στον δημόσιο τομέα, στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και καταλήγουμε στα δικά μας συμπεράσματα και με βάση αυτά υποβάλλουμε προτάσεις προς το Συμβούλιο. Οι δραστηριότητες, ε, οι οίκοι αξιολόγηση είναι πράγματι ιδιωτικέ εταιρείε, αλλά επηρεάζουν πολύ τις χρηματαγορές. Αυτό δεν αποτελεί ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, στο ίδιο θέμα, πρώτο ο κύριος Μέσερ Σμιτ για 30 δευτερόλεπτα. Er Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μας απασχολεί όλους το τι μπορεί να γίνει για να λύσουμε τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Είδα ότι εμφανιστήκατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, πριν λίγες μέρες κύριε Επίτροπε και υποβάλατε την πρόταση τα κράτη-μέλη στο μέλλον να υποβάλουν τις προτάσεις προϋπολογισμού στην Κομισιόν πριν εξετάσουν τα εθνικά κοινοβούλια και συζητήσουν και υιοθετήσουν τις, ε, τα σχέδια προπολογισμού. Μπορείτε παρακαλώ να βαθύνετε σε αυτό το γεγονός δηλαδή ότι η Κομισιόν θα πρέπει στο μέλλον να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους, ε, να πάρει θέση ως προς τους ε, προπολογισμού των κρατών μελών πριν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ για την απάντησή σας. Άκουσα με πολύ προσοχή και τα στοιχεία που μας αναφέρατε και τον τρόπο με τον οποίο μας εξηγήσατε τη στάση της Επιτροπής. Προσπαθώ να καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Αν κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον αντιμετωπίσει μια άλλη χώρα της ευρωζώνης σχετικά προβλήματα με τους οίκους αξιολόγηση και την πίεση των αγορών θα πάμε με αντίστοιχη πεπατημένη; θα υιοθετήσουμε μια λογική βλέποντας και κάνοντας; θεωρούμε ότι με αυτήν την προσέγγιση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα για το πρόβλημα της ελλάδας αντιμετωπίζουμε προβλήματα συνολικά δομικά της ευρωζώνης που κάποια στιγμή ίσως να απασχολήσουν στο μέλλον και άλλα κράτη μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας θυμίσω καταρχήν ότι απαντώ τις ερωτήσεις αυτές στη θέση του Επιτρόπου του κυρίου Ρεν που είναι άρρωστος. Δεν είναι ακριβώς λοιπόν ο χαρτοφυλακάς μου αλλά όσον αφορά τα θέματα εθνικού προϋπολογισμού, τα συζητήσαμε στο σώμα της Επιτροπής πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την παρακολούθηση στο μέλλον και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν αλλά είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Πρόκειται απλά για συζήτηση Ε, για να διασφαλιστεί η επαρκή συζήτηση του θέματος στο Σώμα των Επιτρόπων. Και ο αρμόδιος Επίτροπος θα υποβάλει σχετικές προτάσεις σύντομα και θα μπορέσετε να συζητήσετε το θέμα απευθείας με αυτούς. Η δεύτερη ερώτηση. Δεν υπάρχει λόγος η Κομισιόν να πάρει διαφορετική θέση απέναντι στην Ελλάδα από ότι απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Ελπίζω λοιπόν να μην συνεχίσετε να θέτετε τέτοιες ερωτήσεις προς εμάς, αλλά αν, τις, αν μας ξαναρωτήσετε η απάντηση θα είναι η ίδια την Επίτροπο την κυρία Νέλη Κρούς. Ε, η ερώτηση έχει υποβληθεί από τον κύριο Κρόλη, ερώτηση 30. Εκπροσωπείται, αντιπροσωπεύεται από τον ε, κύριο Έιλουαρντ. Ε, κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο για την απάντηση. Thank you, Mr. President. Το κύριε Πρόεδρε. Σε ένα κόσμο ο οποίος σήμερα προχωρεί γρήγορα τον ε, ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε τις ε, κατάλληλες δομές για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αύριο. Το Μάρτιο 2009 το Συμβούλιο καθόρισε έναν ενδεικτικό στόχο ώστε να έχουμε μέχρι το 2013 κάλυψη 100%. Η στρατηγική 2020 επίσης έθεσε ε, τον πύχη ακόμη πιο ψηλά για το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας για όλους τους Ευρωπαίους 30 MB και για 50% κάλυψη των νοικοκυριών. Η ψηφιακή μέσα στην Ευρώπη που ήταν μία από τις κύριες πρωτοβουλίες της στρατηγικής 2020 θεσπίζει στρατηγική για να προωθηθεί το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε όλη την Ευρώπη και προβλέπεται η οθέτηση αυτού του θέματος σε λίγο καιρό. Θα έχουμε τρία σχετικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρονται ε, τα στοιχεία που αφορούν το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, ε, την πρόσβαση στην ε, τεχνολογίες νέα γενιάς για να έχουμε τη νομική βάση που θα μας επιτρέψει να κάνουμε επενδύσεις σε θέματα διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και τρίτον η πολιτική ραδιοσύχνοτητων, πράγμα το οποίο είναι μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχουμε για τα Wi-Fi ένα ευρύτατο φάσμα. Οι δράσεις, κύριε Πρόεδρε, για την προώθηση του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, πλαίσια της δικής μας ατζέντα συμπεριλαμβάνουν δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και ε, διάφορες υποδείξεις των κρατών μέλων. Πράγμα που θα μας επιτρέψει να μπορέσουμε να έχουμε και εθνικές στρατιστικές ε, για το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας με ιδιωτικές επενδύσεις που θα θεσπίζουν διάφορα θέματα. Έτσι τα κράτη-μέλη μπορούν, πιστεύω, ότι μπορούν να μειώσουν το κόστος των επενδύσεων και να κάνουν πιο βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι που θα τους επιτρέψει να εστιάσουν και την προσοχή τους στο γεγονός ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τους απαραίτητους πόρους ε, που μπορούν ε, μέσω δημοσίων ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων να βελτίσουν. Εμείς προσπαθούμε να ε, αυξήσουμε και τις ιδιωτικές και τις ε, δημόσιες επενδύσεις για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις στόχες μας. Και οι προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν θα πρέπει να γίνουν και στον οικονομικό τομέα ώστε να μπορέσουν εκεί που υπάρχουν μεγάλες διαφορές να τις αμβλύνουμε. Ευχαριστώ. Uh, Κύριος Έλουαρντ, για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ την Επίτροπο για την απάντησή της. Δεδομένου ότι ζούμε σε έναν όλο και περισσότερο ψηφιακό κόσμο, όπως και εσείς αναγνωρίσετε, και αυτό είναι και δεδομένου ότι καθημερινά δουλεύουμε online, μία ομάδα την οποία αφήσαμε κατά μέρο είναι οι γυρεότεροι, οι οποίοι πολλέ φορέ δεν έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία. Τι κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα του αποκλείσουμε από την κοινωνία μα και τι μπορούμε να κάνουμε για να του βοηθήσουμε. Mr. President, ε, Πρόεδρε, όχι μόνο η Κομισιό, αλλά και το Συμβούλιο πήρε την σοφή απόφαση να έχει έναν ενδεικτικό στόχο κάλυψης 100% το 2013 σε όλες χώρες. Δηλαδή 100% σημαίνει 100% θα καλυφθούν οι πάντες και τα πάντα. Έχουμε δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι από τον κύριο Χάρμπορ για 30 δευτερόλεπτα. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω το ερώτηση του κυρίου Κράλλη και με Πρέπει να πω ότι στην Ιρλανδία προβλέπεται ασύρματη πρόσβαση στις νέες αυτές τεχνολογίες του ε, διαδικτύου για όλους. Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως και με θέματα πόρων και περικοπής πόρων που προβλέπονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προσπαθούν όλοι και με την ε, ε, με το δημόσιο να βοηθήσουν την ε, επενδύσεις που θα κάνει και ο δικός τομέας. Αλλά εδώ εφαρμόζονται άλλα κριτήρια. Θα μπορούσαν να δοθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ώστε να μπορέσουν τέτοιου είδους συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την κάλυψη. Ευχαριστώ. Κύριε Τσικάου. Περιμένετε κύριε Επίτροπο και δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης της Οικοσομίας προβλέπει ένα δις ευρώ για την κάλυψη των υποδομών διαδικτύου βρίσκοντας 100%. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε αν μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η κάλυψη. I'm grateful for Είμαι ευγνώμη την πρώτη ερώτηση που μου έγινε κύριε Πρόεδρε. Σωστά. Αναφέρθηκε όταν μιλούμε για το διαδίκτυο και τις οπτικές ίνες, μιλούμε και για το Wi-Fi, για το ασύρματο, για τους... Κάλυψη αυτή 100% την οποία αναφέρουμε γενικά και δεν λέμε με ποιο τρόπο θα καλύψουμε το πρόβλημα όντες. Τώρα, πρέπει να πω ότι εγώ είμαι πολύ θετική για την Ιρλανδία. Διότι όταν υπήρχε δυνατότητα κάλυψης κάποιων δαπανών από τους κοινοτικούς πόρους, από τα διαρθρωτικά ταμεία, πρέπει να πω ότι όντως ε, οποφελήθηκε η Ιρλανδία από αυτή την ε, ευκαιρία που είχε, ε, κάλυψε τη συγχρηματότηση από ποσοστό κάπως λιγότερο 50% σε σχέση με άλλες χώρες που χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους κονδύλια κατά 30% ή δεν έκαναν επενδύσεις καθόλου σε τέτοιου είδους ε, έργα υποδομής. Και πρέπει να πω ότι είναι κάτι το πολύ θετικό, δεδομένου ότι βοηθά την οικονομία να ανακάμψει και δημιουργεί και θέσεις απασχόλησης. Και εγώ βασιζόμενοι στην προηγούμενη εμπειρία, στο που είχαμε το προηγούμενο χαρτοφυλάκιό μου, πρέπει να πω ότι έκανα να κάποιον ε, κανόνων που υπήρχαν για τις κρατικές ενισχύσεις και κάποιες από αυτές αφορούσαν το διαδίκτυο εβραίος φάσματος. Και τι κάναμε, προσπαθήσαμε να δίδουμε περισσότερες συμβουλές και να βοηθούμε τους υπεύθυνους να παίρνουν τέτοιου αποφάσεις που θα τους βοηθούσαν. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να χορηγήσει κάποια κονδύλια συμπληρωματικά. Είναι το σαφές ότι όταν θα, με την αναθεώρηση των κανόνων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις όλοι ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Εάν ε, θέλετε συμβουλές. Αν υπάρχει κάποιο ερωτηματικό, κάποια βεβαιότητα, απευθυνθείτε στον κύριο Αλμούνια, διότι πραγματικά πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όντως κάνει τη διαφορά για τέτοιου είδου θέματα. Και βεβαίως όλα εξαρτώνται από το κάθε κράτος μέλος οριστά. Πιστεύω και επαναλαμβάνω ότι με την ε, κάλυψη 100% όντως κάνουμε κάτι το πάρα πολύ καλό τελικά με τα 100 MB. Ξέρω ότι είναι 100 MB και κατά την άποψή μου πρόκειται για ένα τρομερό βήμα προς τα μπρος. In this uh, debate, our attention is really... Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ελπίζω ότι θα υπάρξει και περαιτέρω πρόεδρος πριν και από το 2001. Τώρα συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις προς τον κύριο Ρεν που εκπροσωπείται από τον κύριο Ντεγκούτ. Η επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση 33 Υποβληθήσα ε, από τον ε, κύριο Πόσελτ. Ε, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για την απάντηση. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα οικονομικά ωφέλη υιοθέτηση του ευρώ ε, έχουν να κάνουν ε, ε, και με τα κρατη αλλά και με το σύνολο της Ευρωζώνης. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ε, έκθεση EMU Aten, ε, μια έκθεση του 2008. Όλα τα νέα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ε, προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ όταν πληρούν τα κριτήρια. Η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, έχουν ρήτρα εξαίρεση για να παραμείνουν εκτό τη ζώνη του ευρώ. Εάν η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσουν να κάνουν αίτηση για προσχώρηση στην Ευρωζώνη, θα ε, αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης ε, ε, επίσης όλους με τους άλλους υποψηφίους. Όπως και στις άλλες περιπτώσεις χωρών που προσχώρησαν στην Ευρωζώνη, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις προσπάθειες. Η Σουηδία δεν έχει τέτοια ρήτρα opt-out, ρήτρα εξαίρεσης. Η Σουηδία δεν πληρεί τα κριτήρια εισαγωγής του ευρώ. Συγκεκριμένα δεν συμμετέχει στον μηχανισμό ε, ισοτιμίας και θα πρέπει να προσαρμοστεί και η νομοθεσία της που αφορά την Κεντρική Τράπεζα. Ε, ωστόσο, η Κομισιόν θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη αυτά που δεν πληρούν τα ε, κριτήρια του ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να τα πληρούν. Κύριε Επίτροπε, δύο συμπληρωματικές ε, ερωτήσεις. Η Κομισιόν δεν θα προσπαθήσει να ενθαρρύνει την Σουηδία να πληρεί τα κριτήρια. Η ε, Σουηδία ε, δεσμεύεται λόγω της σύμβασης. Και τι πιστεύετε για την Εσθονία. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει στο εγγύς μέλλον να προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, σωστά αναφέρθηκε, η Σουηδία δεν πήρε τα κριτήρια. Ε, ανέφερα τα δύο κριτήρια. Το ένα είναι ότι δεν συμμετέχει στο μηχανισμό ισοτιμίας και κάποια στοιχεία της νομοθεσίας για την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας θα πρέπει να ε, προσαρμοστεί στην συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Τα κριτήρια αυτά είναι δυνατόν να αλλάξουν, δεν είναι οικονομικά κριτήρια. Δεν έχουν να κάνουν με το χρέος ή το έλλειμμα. Εγώ προτείνω να ρωτήσετε τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Ρεν, ε, για το αν η ε, Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει δράση. Ε, ο κύριος Ρεν δυστυχώς είναι άρρωστος όσον αφορά την Εστονία, από ό,τι γνωρίζω. εξετάζονται ακόμα τα κριτήρια σύγκληση και δεν υπάρχει οριστική θέση της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για την απάντηση. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στην ερώτηση 34. Excuse me. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Οι δείκτες αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπήρξε μια αποσύνδεση ανάμεσα στα ποσοστά ανάπτυξης και τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Αυτό οδήγησε ε, σε ε, ανταγωνιστικό ε, ε, μειονέκτημα το οποίο, ανταγων... Ε, το οποίο κατοπτρίζεται στο ολένα και φαινόμενο έλλειμμα καθώς και στις χαμηλότερες εξαγωγές. Υπήρξε ένα μεγάλο κόστος, εργατικό κόστος. Τα, τα τελευταία χρόνια η οικονομική ανάπτυξη βασικά οδηγήθηκε, καθοδηγήθηκε από τις μεγάλες ε, κρατικές επενδύσεις. 80% αυξήθηκαν οι κατακεφαλήν δαπάνες. Αυτό το πρότυπο φυσικά δεν ήταν δυνατό να σταθεί. Αυτό σήμαινε μεγάλο έλλειμμα για την κυβέρνηση, για το κρατικό έλλειμμα και αυξημένες ε, μικροδαπάνες ε, και μεγάλες ε, ανισορροπίες όσον αφορά το εξωτερικό χρέος. Αυτό οδήγησε στο ότι ο δημόσιος τομέας απορρόφησε το τελευταίο τμήμα της, ε, ε, διαθέσιμης χρηματοδότησης και ο ιδιωτικός τομέας επλήγει καθώς και ε, επηρεάστηκαν αρνητικά οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Τα μέτρα λιτότητας είναι λοιπόν απαραίτητα ώστε η ελληνική οικονομία να ξεκινήσει σε, μια, σε νέα θεμέλια ισχυρότερα και να πετύχει την οικονομική παγίωση. Η Κομισιόν ορίζει πως τα μέτρα αυστηρότητας καθώς και η, μετρίαση των ημερομεστίων μπορεί να έχει επίπτωση στην ζήτηση, αλλά αυτά τα, αυτά τα μέτρα θεωρούνται απαραίτητα ώστε να τεθούν τα θεμέλια για πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξη για την ευρωπαϊκή, ελληνική οικονομία μακροπρόθεσμα. Η Ελλάδα υιοθέτησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει το έλλειμμά τη και για να ανορθώσει και πάλι την οικονομία τη. Τα μέτρα παγίωση που έλαβε η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικά ώστε να, να στηριχθεί η βιωσιμότητα και έχουν στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από το Διεθνές Μαζικό Ταμείο. Τα θαραλέα μέτρα αυτά που περιλαμβάνονται στα πακέτα που ανακοινώθηκαν το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2010 συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τις προβλεπόμενες ε, περικοπές μισθών μέσω του περιορισμού των επιδομάτων καθώς και το χριστουγεννιάτικο και πασχαλινού δώρου των ε, υπαλλήλων αλλά και μέσω της ε, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Το, 2000, το Μάρτιο του 2010 η Κομισιόν ε, κατέληξε στο ότι η Ελλάδα εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2010 μέσω των μέτρων που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί να διασφαλιστούν και να επιτευχθούν οι στόχοι δημοσιονομικοί για το 2010. με τελευταία της ανακοίνωση κύριε επίτροπε η ελληνική στατιστική αρχή νομίζω αυτό έγινε σήμερα ε, ότι η ανεργία στην ελλάδα σκαρφάλωσε στο 11,3 από τους οποίους ανέργους σχεδόν η μισή το 45% είναι νέοι έως 34 ετών. Στις δε ηλικίες από 25 μέχρι 34, 14,6 είναι η ανεργία, στις πιο παραγωγικές δηλαδή ε, ηλικίες και σημειώνω ότι αυτή η γενιά των νέων ανθρώπων στην ελλάδα αμείβεται με ιδιαίτερα χαμηλού μισθού πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι η γενιά των 700 ευρώ που λέμε στην ελλάδα φοβόμαστε ότι θα πάει ακόμη παρακάτω πλέον. πρέπει να είμαστε λοιπόν νομίζω προσεκτικοί σε αυτέ τι γενικεύσει ειδικά σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την ανεργία γιατί αντιλαμβάνεστε η ελληνική κοινωνία ανησυχεί. θεωρείτε λοιπόν ότι ενώ υπάρχει αυτή η ανεργία στην ελλάδα όλα αυτά τα προβλήματα στην ελλάδα με περικοπές και νέες απολύσεις μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Κύριε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά και ανησυχούμε πολύ με την, ε, για την ανεργία στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως από την άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικό ε, οι βασικές ε, συνιστώσεις της οικονομίας να γίνονται σεβαστές και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα τα, ε, οι μισθοί όταν ανεβαίνουν περισσότερο από την παραγωγικότητα έχουμε πρόβλημα και βασικά αυτό είναι που συνέβη στην Ελλάδα αλλά συνειδητοποιώ πως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ιδιαίτερα για τους νέους και Φυσικά και παρακολουθούμε την κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να αντιδράσει και το κράτος μέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι επί της αρχής. Με αφορμή την ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος, ο συνάδελφος στη γραπτή. Λέει ο εκπρόσωπος του κυρίου Ρεν προφανώς πιθανολόγησε ότι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γίνουν περικοπές στην Ελλάδα η ερώτηση κύριε επίτροπε είναι με ποιο δικαίωμα επιτηρητές της κομισιόν εκπρόσωποι επιτρόπων και ενδεχομένως επίτροποι μιλούν πιθανολογούν προβλέπουν πιέζουν τι πρέπει να κάνει η ελλάδα σε τομείς που δεν αφορά την κοινοτική πολιτική αλλά που αφορούν την εθνική πολιτική όπως είναι τα θέματα μισθών συντάξεων δημόσιας διοίκηση υγείας ποιος νομιμοποιεί αυτές τις δηλώσεις από πού αντλούν αυτή την αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία να ρωτάνε ή να επιδιώκουν ή να πιθανολογούν τέτοιες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο. Thank um, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά, δεν ζητάμε να μειωθεί η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Όχι. Η ανεργία αυξάνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ένα μεγάλο κομμάτι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσμα της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να να κάψει η ελληνική οικονομία αν θέλουμε αυτή να επιβιώσει και μακροπρόθεσμα. Ε, και επίσης θέλουμε να διαπροστατεύσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση που είναι τεράστια σημασία για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό λέμε. Σίγουρα πάντως δεν λέμε πώς θα πρέπει να αυξηθεί η ενεργία. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα δυστυχώς. Είναι μια συνέπεια πολιτικών που έχουν ε, ακολουθηθεί ε, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 35 έχει υποβληθεί από τον ε, κύριο Κόζα, εκπροσωπείται από την κυρία Γκάλ. Ε, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για την απάντηση. Number 35. Thank you, uh, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν έπληξε το φθινόπωρο 2008 η οικονομική κρίση την Ουγγαρία, προσπαθήσαμε με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης με 6,5 ευρώ να μπορέσουμε να προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε. Και έφτασε το ποσό αυτό στα 20 δις ευρώ με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Θα ήθελα να πω ότι αυτή, χωρίς αυτή την ενίσχυση η Ουγγαρία θα είχε πολύ περισσότερα προβλήματα στην οικονομία της από το 6% ε, μείωση που είχε πέρσι του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της σταθερότητας φέτος. Εξάλλου, πρέπει να πω ότι αν δεν είχαμε την, δεν υπήρχε δική μας υποστήριξη θα υπήρχαν πολύ περισσότερα προβλήματα και οι, διάφοροι, και οι μύες των δαπανών θα ήταν πολύ περισσότεροι. Πράγμα το οποίο επέτρεψε να υποστηρίξουμε την χρηματοδότηση του ελλείμματος, να μειώσουμε τον αριθμό των ανέργων και να περιορίσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις κρίσης συμπεριλαμβανομένης και των κρίσεων που πήραν για να μπορέσουμε να είμαστε ε, αξιόπιστοι και για να μπορέσουν ε, να πάνε οι επενδυτέ στην Ουγγαρία θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική εκ μέρους της ε, κυβέρνησης και μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας και φορολογικά μέτρα. Βάσει τη αρχή επικουρικότητα είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για τα μέτρα κοινωνική πολιτικής τα οποία θα λάβουν δράσεις της κυβέρνησης και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν για να γίνουν οικονομίες στον κρατικό προϋπολογισμό και καλύτερη στόχευση των δαπανών είναι κάτι το απαραίτητο. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, és köszönöm a választ. Kósa képviselő úr eh, eh,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 jön itt létre erről kérdezném a véleményét. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι, όπως ξέρετε, υπεύθυνο για αυτό το φάκελο στην Κομισιόν, αλλά μου φαίνεται ότι αναφέρεται στο πακέτο των 100 ε, δις ε, η κυρία Βουλευτής. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο προήλθε από το δι Ταφ και δημιούργησε μετά ένα έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας σας. Βεβαίως, τα 20 δις είναι κάτι το οποίο δόθηκε ως συμπληρωματική βοήθεια και το κράτος σας έπρεπε να πάρει μέτρα για να ξεπεράσει την κρίση, αλλά το ποσό αυτό δεν δόθηκε σε αυτό το χώρο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, η απάντηση που δώσατε κατά την άποψή μου δεν παρακολουθεί την προβληματική και τον προβληματισμό της ε, ερώτησης. Και με αφορμή την υπόθεση της Ελλάδας θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σας έχει προβληματίσει καθόλου η είσοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ένα εξωτερικού οργανισμού, στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πήγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έσπηρε την καταστροφή θα έλεγε κανείς. Η ερώτηση λοιπόν είναι, έχει προβληματίσει την Κομισιόν γιατί μπήκε το διεθνές νομισματικό ταμείο στην ευρωπαϊκή ένωση και η πιο ερώτηση σε ποια συνθήκη σε ποιο άρθρο προβλέπεται η συμμετοχή του διεθνούς νομισματικού ταμείου στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ένωσης. γιατί δεν επιλέγει μια ευρωπαϊκή λύση για την περίπτωση της ελλάδας που προβλέπουν οι συνθήκες στο άρθρο 122 παράγραφο 2. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε uh, uh, Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Εάν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ χρειαστεί να παρέμβει στην Ελλάδα, θα γίνει αιτήση της Ελλάδος αυτό. Και όπως ξέρετε, υπήρξε ευρωπαϊκή ε, απόφαση στο Eurogroup να μπορέσει να βοηθηθεί αν χρειαστεί ένα κράτος μέλος και να βοηθηθεί από το Δέλτα Νιτάφ. Αλλά μόνο αυτό θα γίνει αυτό μόνο αν υπάρχει έτοιμα εκ μέρους της ε, ενδιαφερόμενης χώρας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι εκρεμές προς το παρόν. Συζητείτε ακόμη. Ε, της κυρίας ε, Ελένης ε, Θεοχάρους. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο για την απάντηση. where's the answer? Well, uh... Uh, Κύριε Πρόεδρε, Ναι, ναι, το βρήκα. Να σας ζητήσω, παρακαλώ, μήπως να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, γιατί εγώ αντικαθιστώ τον κύριο Ρέν. Και κανονικά η ώρα των ερωτήσεων να σταματά στις 8 και έχω μια άλλη ενηλυμένη υποχρέωση. Thank you. No, I have no time. I cannot stay. Δεν έχω χρόνο, δεν μπορώ να μείνω. Πρόκειται... Δεν δέχομαι, δεν δέχομαι πως δεν έχετε χρόνο. Άμα δεν έχετε χρόνο, κοιτάξτε εδώ. Εδώ ε, έχω πολλές δεσμεύσεις, επίσης ανελημμένες υποχρεώσεις και έχω κάτσει εδώ να... τόση ώρα περιμένω να έρθει η ερώτησή μου. Ενώ απαντήθηκαν ένα σώρο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Παρακαλώ, ε, να είστε ευγενικό απέναντί μας. Είναι πραγματικά υπεροπτικό απέναντί μας να λέτε πως δεν έχετε χρόνο. Κοιτάξτε, εξαρτάται από τον Πρόεδρο να αποφασίσει, αλλά... Δεν απαντώ, δεν απαντώ σε ερωτήσει που έχουν υποβληθεί σε μένα, αλλά αντικαθιστώ τον κύριο Ρεν γιατί είναι, είναι ασθενή. Δεν μπορεί να είναι εδώ. Θα πρέπει αυτά να τα πείτε στον πρόεδρο. Εγώ α, σέβομαι την ε, κυριαρχία του προέδρου εδώ. Έχετε δίκιο, γιατί τονίζετε ένα πρόβλημα. Εσεί την καθιστάτε τον Επίτροπο Ρεν, πράγμα που είναι βέβαια ατυχέ δεδομένων των, ε, δεδομένων τη σημασία των ερωτήσεων. Ωστόσο, μέχρι τι 8.30 προβλέπεται η ώρα των ερωτήσεων στο πρόγραμμά μα. Και δεδομένων των συνθήκων, δεν μπορώ βέβαια να σα δέσω εκεί στην καρέκλα, αλλά μπορώ να σα πω ότι αυτό που αναμέναμε ήταν αφού εσείς ε, είχατε την ατυχία να για τον κύριο Ρεν, οφείλετε να το καταστήσετε πλήρως για όλες τις ερωτήσεις. Οπότε παρακαλώ προχωρήστε και απαντήστε στην κυρία Θεοχάρους. Δεν είχα καταλάβει πως θα καθυστερούσε η ώρα των ερωτήσεων, αλλά όπως είπα ήδη, εσείς έχετε την Προεδρία και εσείς ε, αποφασίζετε τι θα κάνω, οπότε θα συνεχίσω. Και ό,τι γίνει έγινε. Η κρίση την οποία διανύουμε ήταν η χειρότερη με τα πολεμικά και στήχησε πολύ στην παγκόσμια οικονομία και σε αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις χώρες ε, της Ευρωζώνης. Αυτό φυσικά έχει επηρεάσει και την Κύπρο που είναι μια πολύ μικρή ανοιχτή οικονομία. Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις που έχουν ε, ε, εκδοθεί από την ε, Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, φαίνεται ότι η ανάπτυξη έχει μειωθεί κατά 1,7% το 2001. Είναι η πρώτη φορά όπου καταγράφεται αρνητικό ποσοστό μεγέθυνση στα τελευταία 25 χρόνια στην Κύπρο. Αυτά συνδυάζονται με την άνθηση των, ε, ε, της αγοραστικής της, της αγοράς ακινήτων και με την πρόσφατη τροποποίηση των στοιχείων EDP που μετέδωσαν τα, η Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία και αξιολογούνται τώρα από την Eurostat. 6,1 της, ε, του ΑΕΠ είναι το, φαίνεται να είναι το κρατικό έλλειμμα και θα έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2009. Η υπηρεσία της Κομισιόν ε, υπεύθυνη για το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης είναι έτοιμη να ετοιμάσει τη σχετική έκθεση μόλις θα έχουν ε, ολοκληρωθεί τα στοιχεία. Μόλις θα είναι έτοιμη αυτή η έκθεση θα αποφαστεί από το Συμβούλιο αν το έλλειμμα είναι υπερβολικό και σε τέτοια περίπτωση το Συμβούλιο θα προβεί σε συστάσεις στην Κύπρο ε, και θα καθεσπίσει προθεσμίες ώστε να αναλυθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ η Κύπρος έχει υποβάλει το, το πρόγραμμα σταθερότητάς της που φτάνει μέχρι το 2013 και αυτή τη στιγμή η Κομισιόν αξιολογεί την ενημέρωση του προγράμματος σταθερότητας της Κύπρου και θα ενημερώσει και το Συμβούλιο ώστε αυτό να λάβει θέση. κύριε Επίτροπε, θα ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό αν δεν δίνατε απάντηση από τη στιγμή που η ερώτηση ετέθηκε. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να μου πείτε αν η Κύπρος κινδυνεύει να τεθεί υπό επιτήρηση και αν είστε ικανοποιημένο από το πρόγραμμα σύγκλησης. Βεβαίως, κάτι είπατε ότι αξιολογείται, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν είστε ικανοποιημένο από το πρόγραμμα σύγκλησης που υπέβαλε η κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτά που είπα. Ότι δηλαδή θα γίνει η αξιολόγηση είναι η φυσιολογική διαδικασία που εφαρμόζεται για όλα τα κράτη-μέλη, άρα και για την Κύπρο. Αν η Κομισιόν καταλήξει ότι πρόκειται για υπερβολικό έλλειμμα, τότε θα ε, προβεί σε σύσταση, σε συστάσεις προς την Κύπρο. Επόμενη ερώτηση, ερώτηση νούμερο 37, από τον κύριο Μέσερ Σμιτ. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ για την απάντησή σας. Number 37. Υπαριθμό 37. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο αξιότιμος κύριος Βουλευτής ε, φαίνεται να θεωρεί ότι η ανεξάρτητη οικονομική πολιτική στην Ελλάδα θα ήταν τρόπος να ε, ανακουφιστεί η κρίση που ε, πλήττει τη χώρα. Αυτό δεν είναι σωστό. Τα υψηλά επιτόκια στις στα ελληνικά δάνεια έχουν να κάνουν με ιστορικούς παράγοντες. Οι ε, ελληνικές τράπεζες ε, παρέχουν ε, αρκετή ρευστότητα και στην Ευρώπη και, στους ελληνικούς, και στα ελληνικά πιστοτικά ιδρύματα. Ωστόσο, απαιτείται ένα σύστημα κειμενόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών και όπως φαίνεται στις εκθέσεις της Επιτροπής στην έκθεση του, ε, της Επιτροπής του 2008 η προσαρμογή στην Ευρωζώνη δεν ήταν ομαλή στο παρελθόν και γι' αυτό η Επιτροπή προτείνει διαδικασία επιτήρησης για να ε, εντοπιστούν και να, και να αντιμετωπιστούν ε, αδυναμίες στα κράτη-μέλη. Ε, απάντησα και σε προηγούμενες ερωτήσεις πάνω στο σχετικό θέμα. Ε, ναι, υπάρχουν πολλές δυνατότητες να ρυθμίσει κανείς το συνάλλαγμά του, εάν έχει κανείς την ανεξαρτησία του. Ε, τα μέλη του ευρώ δεν έχουν την ανεξαρτησία αυτή, διότι έχουν βάλει στα χέρια της Φραγκφούρτης ε, πολλά μέσα που είχαν στο παρελθόν και δεν είναι αλήθεια ότι τα επιτόκια δεν διαφέρουν ε, εντός της ε, Ευρωζώνης. Για παράδειγμα, τα επιτόκια στα ελληνικά ομόλογα είναι πολύ πιο ψηλό από ότι το δανέζικο. Θέλω η Επιτροπή να ομολογήσει ότι αν η Ελλάδα δεν ήταν κλειδωμένη στην θέση που ε, υπαγορεύει η Φραγκφούρτη, η ε, Ελλάδα θα είχε υποτιμήσει το ε, συνάλλαγμά της και αυτό θα είχε ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα. Ε, κύριε Βουλευτά, σίγουρα όχι. Η ιδέα της νομισματικής ένωσης είναι ότι ο καθένας γνωρίζει ότι όταν γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ε, ότι δεν μπορεί πια να ε, υποτιμήσει το συνάλλαγμα διότι δεν υπάρχει πια ελληνικό συνάλλαγμα. Οι Έλληνες έχουν ως συνάλλαγμα δικό τους το ευρώ. Η ανατίμηση λοιπόν αντίκειται στην η ιδέα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και η Ελλάδα δεν ε, είναι τυχαία μέλος της ε, Ευρωζώνης, πληρεί όλα τα κριτήρια, πραγματικά όλα τα κριτήρια. Κύριο ε, Γκέι Μίτσελ, έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε για την απάντηση. Number 38. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απέδειξε η κρίση ότι χρειάζεται να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο επίλυσης κρίσεων στην Ευρώπη. Ένα θέμα, το, ένα από τα θέματα είναι με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε μέσω των ε, των Ιδρυμάτων και των θεσμικών οργάνων που έχουμε το θέμα αυτό και αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκε το σχετικό συμβούλιο. Το θέμα της ε, δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο όταν έχουμε επίγουσες καταστάσεις ε, οικονομικής ε, ενίσχυσης κάποιου. Παρ' όλα αυτό δεν χρειάζεται νέος χρονισμός για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Εμείς αναλύουμε τις προτάσεις, έχουν αναλυφθεί κάποιες δεσμεύσεις και θα πρέπει να αναλυφθούν από όλα τα κράτη-μέλη που είναι μέλη της ε, ΟΝΕ για να μπορέσει να συνεχίσει να ισχύει το σύστημα και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός για όλες τις ενέργειες που γίνονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στον Επίτροπο. Πρέπει να πω ότι είμαστε όλοι κάπως εκτευρισμένοι γιατί πολλοί από εμάς δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε στις οικογένειές μας. Με την απάντησή του θα ήθελα να πω το εξή τον Επίτροπο. Μιλήσατε για μεσοπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό για σας. Ένα χρόνο, 18 μήνες για να μπορέσετε σε τέτοιου είδους θέματα να δώσετε μια πιο συγκεκριμένη και οριστική απάντηση. Την ερώτηση για το πλαίσιο αυτό το μακροτόπιο θα πρέπει να την κάνετε στον κύριο Ρέιν. Αν δείτε τις συστάσεις που κάναμε και τη συμφωνία η οποία επιτεύθηκε για να υποστηριχθεί κυρίως η Ελλάδα συνδυάζοντας ε, διμερή δάνεια και υποστήριξη από το ΔΕΛΤΑ θα δείτε ότι είναι σαφές ότι η Κομισιόν είναι υπέρ τη άποψης ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα δεν μπορεί να επιληθεί με την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, γιατί αυτό θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο από ό,τι χρειαζόμαστε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για σχέδια μακροπρο... μέσω πρόθεσμα, τα οποία βλέπουμε θετικά, αλλά σε σχέση με ένα με το ειδικό χρονοδιάγραμμα που θα χρειαστούμε, παρακαλώ κάντε την σχετική ερώτηση στον Επίτροπο Ρέν. Η τελευταία ερώτηση είναι από την κυρία Κράτσα, η ερώτηση 39. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για την απάντηση. Uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν μακρόν ε, υποστήριζε την ε, εις οικονομική εποπτεία. Αυτή, η σημασία αυτού αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δήλωση για την, την Ευρωζώνη και τη δημόσια οικονομία. Η Κομισιόν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πλήρως τη νέα συνθήκη για ισχυρότερο συντονισμό και καλύτερη διακυβέρνηση. Θα υποβάλουμε προτάσεις ώστε να πλαισιώσουμε την ανάπτυξη ενός συνολικού πλαισίου για μια συνολική αντιμετώπιση κρίσεων μέχρι του νέου άρθρου 136 της συνθήκης σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάνει προτάσεις για να ενισχύσουμε την ε, εποπτεία στην Ευρώπη, ε, στην Ευρωζώνη, τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες καθώς και το μηχανισμό επίλυσης κρίσεων για τις χώρες της Ευρωζώνης. Όσον αφορά την Οικονομική Επιτροπή, ενισχυμένη πολιτική για την οικονομική βιωσιμότητα λόγω του αντικτύπου της κρίσεως καθώς και κίνητρα για τη συμμόρφωση προς τις προληπτικές και διορθωτικές διαστάσεις της ε, διόρθωσης. Ε, θα πρέπει βέβαια όλα αυτά να γίνουν εγκαίρως, ε, ώστε να ληφθεί υπόψη βέβαια και η δυνατότητες της κάθε, της κάθε χώρας και των, της οικονομίας αυτής. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις όπου οι κανόνες διαρκώς παραβιάζονται. Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να είναι πιο αποτρεπτικές και τα κίνητρα να ενισχυθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες επιπλέον των φορολογικών είναι πολύ σημαντικό θέμα για την σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Οι αποκλήσει ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ιδιαίτερα για τα κράτη που συνδέονται με το ευρώ, λόγω του μεγάλου βαθμού οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ε, διάχυσης ε, του αντικτύπου των κρίσεων. Υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες μάλλον υπάρχουν μεγαλύτερες, λιγότερες μάλλον δυνατότητες προσαρμογής, οι οποίες κοστίζουν ε, και υπερβολικά πολύ. Είναι όλα αυτά πολύ σοβαρές ανησυχίε όσον αφορά τη λειτουργία της νομισματικής ένωσης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας πρώτης που προηγήθηκε της κρίσης, Δημιουργήθηκαν διάφορες ε, χώρες ανισορροπίες σε διάφορα κράτη-μέλη ε, όπως φούσκες, ε, προβλήματα στις αγορές ακινήτων, αδυναμίες στην εγχώρια ζήτηση σε ορισμένες χώρες πλεονασματικές καθώς και η σώρευση εξωτερικού χρέους, καθώς και η λανθασμένη κατανομή των πόρων που δίνονταν για την προσαρμογή, καθώς και αυξημένη ε, ευαισθησία της δημόσιας οικονομίας. Χώρες που είχαν ε, βασιστεί στα εμπορικά πλεονάσματα αποτέλεσαν τα πρώτα θύματα της ε, κρίσης. Γι' αυτό και η συμπληρώση της υποπτίας της οικονομίας ε, θα είναι αντικείμενο προτάσεων που θα προκύψουν από την ε, Κομισιόν όσον αφορά την Ευρωζώνη, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες, ε, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως τα προβλήματα και να διορθώνονται εγκαίρως αυτά. Η Κομισιόν ε, έχει προβλέψει τον ad hoc μηχανισμό για την ε, βοήθεια προς την Ελλάδα. Αυτό εξυπηρετεί μια ανάμεση ανάγκη, ωστόσο θα πρέπει να δούμε έναν τέτοιο μηχανισμό με μεγαλύτερη ε, και ταχύτερη δυνατότητα ενεργοποίησης με συγκεκριμένους κανόνες αυστηρούς όσον αφορά τη βοήθεια προς μια χώρα της Ευρωζώνης. Οι προτάσεις για την αυξημένη οικονομική εποπτεία και συντονισμό στην Ένωση, στην ε, Ευρωζώνη, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής για το 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή πρέπει να φύγετε, δεν σας διακόψα. Οι διερμηνείς ε, δεν τρελάθηκαν με την ταχύτητα με την οποία μιλήσατε. Δεν μπόρε σαν να αποδώσουν απόλυτα πιστά το κείμενό σας. Πρέπει να καταλάβατε όσο γινόταν και... Για 30 δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε να ρωτήσετε συμπληρωματική ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ε, επιτρέψτε μου να επανέλθω στο θέμα της εποπτείας και της ανισορροπίας ε, αυτό που θέλω ε, με την ερώτησή μου να μάθω είναι εάν θα μας απασχολήσει έστω για πρώτη φορά σοβαρά η απόκληση όχι μόνο οι ανισορροπίες οι δημοσιονομικές αλλά η απόκληση οικονομική και όχι μόνο οι μηχανισμοί εποπτείας για τη δημοσιονομική πειθαρχία αλλά για την αντιμετώπιση των αποκλήσεων. η κρίση η διεθνής η κρίση η ελληνική έφεραν στην επιφάνεια όλες αυτές τις αδυναμίες της ευρωζώνης σας ευχαριστώ πολύ. σημειώνω την αναφορά στο άρθρο 136 είναι πολύ σημαντική η ενεργοποίησή του αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα συντονισμού και πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές αποκλήσεις. σας ευχαριστώ. Ε, ε, ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητώ Ζητήσω συγγνώμη από τους διερμηνείς. Αλλά Πώς καταλαβαίνετε είναι κάπως εξαιρετική η κατάσταση, έκτακτη. Και προσπαθώ να απαντήσω και τις ερωτήσεις μέσα την ώρα των ερωτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 8.30, εν περιπτώσει, σε σχέση με τη συμπληρωματική ερώτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε στην ε, ρίζα της κρίσης στην χώρα σας, που είναι ακριβώς το γεγονός ότι αυτές οι ανισορροπίες έχουν ε, δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Είναι μεγάλο το πρόβλημα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα ε, πολύ και, τις, ε, και το χρέος και αυτό φυσικά είναι θέμα εθνικών πολιτικών καταρχήν. Τώρα, αν είναι καλύτερο να υπάρχει στενότερη παρακολούθηση, η απάντηση είναι ναι. Και γι' αυτό και προτείνουμε και ένα νέο πρόγραμμα γι' αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2002 η Κομισιόν έκανε μια πρόταση ώστε να μπορεί να σταλεί μια ελεγκτική αποστολή για να ελέγξει τα νούμερα. Ε, αυτό δεν έγινε δεκτό από το κράτος μέλος. Αυτό η Κομισιόν ναι γνώριζε πως ε, ο έλεγχος ήταν πάντοτε σημαντικό ώστε να τηρούνται και να είναι συμβατοί οι εθνικοί προπολογισμοί με την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε πίτροπε, κύριε Τεκούτ. Ε, all I can tell you is that Ren... Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα σας χρωστάει μεγάλη χάρη όλη Ρεν εδώ να το χρησιμοποιήσετε αυτό στην επόμενη φορά που θα είσαστε στην ώρα των ερωτήσεων. Οι δεν δόθηκε απάντηση η του χρόνου θα λάβουν γραπτή απάντηση. Η ώρα των ερωτήσεων έληξε. Ε, αναστέλλεται τώρα η συνεδρίαση ως τις 9 η ώρα. Ε, το βράδυ ευχαριστώ πολύ.